για να παρακολουθήσετε τις συζητήσεις μας μέσω διαδικτύου. Έχουμε τα σημεία 4, 5, 6, 7, 8, Τα εξετάσαμε αυτά τα σημεία που ανέφερα Λοιπόν, το, μικρόφωνο, το κάθε μικρόφωνο συνδέεται με την κάμερα. 6, 7, 8, τα εξετάσαμε. Τώρα λοιπόν, καλωσορίζω τους επισκέπτες που καταφθάνουν. Τους ζητώ να κάνουν λίγη ησυχία, να πάνε στις θέσεις τους. διακόπτοντας ε, όσο πιο λίγο γίνεται τις εργασίες μας. Και δίνω το λόγο για το σημείο 10, 11, 12, 13 και 14 το λόγο δίνω στη συνάδελφό μας Μπάρμπαρα Ματέρα. Ευχόμενος ε, το καλώς ήρθε στους ε, επισκέπτες της, στους προσκεκλημένους της. Έχει πολλά σημαντικά σημεία, κινητοποίηση, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Διάφορα σημεία που αφορούν αυτό το θέμα. Η Μπάρμπαρα λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο για να μιλήσω για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Είναι από δύο χώρες το αίτημα, από την Ισπανία και την Πολωνία. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο αργή ε, γιατί μιλάω γρήγορα συνήθω και μου είπαν ότι πρέπει να μιλάω πιο αργά για να διευκολύνω του διαρμηνεί και να μπορούν να, να μεταφράζουν με πιστότητα αυτά που λέω. Λοιπόν, το πρώτο έτοιμο είναι από την Ισπανία. Υποστηρίζει 528 εργαζομένους που απολύθηκαν από 76 εταιρείε στον τομέα των οικοδομών από τι επιχειρήσει ζητήθηκε από υποστήριξη και είναι ένα εκατομμύριο 420 εκατομμύρια 420.000 ευρώ. Η άλλη είναι από την Ισπανία, από την περιοχή της Βαλένθια. Ζητείται υποστήριξη για 350 εργαζομένους που απολύθηκαν από 143 επιχειρήσεις που κινούνται στον τομέα της κρουστεφαντουργίας. Το ποσό που ζητείται είναι 2 εκατομμύρια 60.000 ευρώ περίπου. Το τρίτο αίτημα αυτή τη φορά, και αυτό πάντα από την Ισπανία, από την περιοχή της Αραγώνας, όπου εκεί 1154 απολύσεις σε 593 ε, διάφορες επιχειρήσεις που κινούνται στον τομέα του, της, του λιανικού εμπορίου. Το ποσό που εζητήθηκε είναι 1.560.000 ευρώ περίπου. Τελευταίο αίτημα προέρχεται και αυτό από την Ισπανία. Ζητείται υποστήριξη 508 εργαζομένων τη εταιρεία Automotive που είναι στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και το ποσό που ζητείτε είναι 330.000 ευρώ περίπου. Λοιπόν πάμε στο πιο δύσκολο τμήμα ή να μιλήσουμε για τα δύο πολωνικά αιτήματα, γιατί έχω δύσκολο να διαβάσω τα ονόματα των εταιριών, να τα προσπαθήσω. Πρώτο αίτημα ζητά υποστήριξη για 590 εργαζομένους της εταιρείας Wilkol Polski Automotive του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ζητείται μια υποστήριξη 630.000 ευρώ. Το δεύτερο αίτημα είναι υποστήριξη 189 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία, πιο δύσκολο το όνομα εδώ, Τσετζιέλσκι Πόσναν, που κινείται στον τομέα της ναυτιλίας. 115.000 ευρώ περίπου ζητούνται εδώ. Επενθυμίζω εδώ ότι αυτά τα αιτήματα θα ψηφιστούν το Δεκέμβριο και όσον αφορά την Επιτροπή Υπηρεπολογισμών, και όσον αφορά την Ολομέλεια. Σήμερα πιστεύω, αν μου το επιβεβαιώσει ο Πρόεδρος, ψηφίσουμε δύο αιτήματα τα οποία ήδη παρουσίασα την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τη γερμανική περίπτωση και την σλοβακική που ήδη παρουσίασα κατά το παρελθόν. Και εδώ κλείνω. Ήθελα να σας μιλήσω για δύο τροπολογίες που μου πρότειναν δύο συνάδελφοι και λυπούμε που απουσιάζουν, Άλβαρο και Άουγκλαντ, που είναι υπέρ Είμαι υπέρ της πρώτης τροπολογίας όπου ζητείται η επανεισαγωγή, η επανένταξη των απολυμένων στον επαγγελματικό ιστό να έχουν μια θέση εργασίας υπό διαφορετικές συνθήκες αλλά μέσω μακρά μακράς διαρκείας συμβάσεις. Είμαι υπέρ αυτής της ε, προτάσεως ε, που είναι κοντά σε αιτήματα των εργαζομένων. Εγώ δεν είμαι υπέρ όμω τη τροπολογία υπαριθμών 2 που υπευλήθη από τους ίδιους συντάκτε Άλβαρο και Άγκλαντ ε, διότι ε, οι τροπολογίες αυτές υπογραμμίζουν τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Παγκοσμιοποιήσεως και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τομέα. Υπογραμμίζουν τον αριθμό των ετοιμάτων που αυξάνεται όσον αφορά το Ταμείο τη παγκοσμιοποίηση και από αυτό συνεπάγεται, συμπεραίνονται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών γίνεται κακή χρήση ε, των διαθροτικών ταμείων. κακή η έλλειψη χρήσεως των διαθροτικών ταμείων. Στους δύο συναδέλφους που δεν είναι εδώ σήμερα θα ήθελα να πω ότι αληθεύει ότι υπάρχει συμπληρωματικότητα όσον αφορά τι δράσει που χρηματοδοτούνται από τα δύο ταμεία, αλλά μιλάμε όμω ταυτόχρονα για δύο ταμεία που είναι εντελώ διαφορετικά. Διότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπω γνωρίζουμε, είναι ένα ταμείο διαθροτικό, ε, πολύ πιο άκαμπτο και αργό όσον αφορά τι διαδικασίε. Το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης που πρόσφατα δημιουργήθηκε, που είναι ένα ταμείο πιο ευέλικτο, πιο γρήγορο και πιο εύκαμπτο, είναι ένα ταμείο που έχει σαν στόχο να δώσει υποστήριξη κατά περίπτωση στους εργαζομένους που απολύονται. λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για συμπληρωματικότητα αυτών των δύο ταμείων. Όμως, θέλω να πω ότι δεν είμαι υπέρ της τροπολογίας, λοιπόν, για όλα αυτά που είπα, δεν είμαι υπέρ της τροπολογίας υπαριθμών 2 και ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ συνάδελφοι, συγχαρητήρια που μπορέσετε και να μας παρουσιάσετε τόσο σαφώς και συνθετικά. Τα euh, διάφορα σχέδια. Τρία ισπανικά, ένα πολωνικό, δύο πολωνικά μάλλον. Να το οποίο τα είπα η συζήτηση σήμερα χωρίς πληροφορία και μετά τα θέματα που θα ακολουθούν από ψηφοφορία. Ένα από τη Σλοβενία και ένα από τη Γερμανία. Και να μας παρουσίασαν τις απόψεις σας για τις δύο πληγές που έχουν υποβληθεί. Θα ήθελε κάποιο το λόγο για την κοινή συζήτηση αυτών των διαφόρων σχεδίων. Όχι. Ωραία. Θαυμάσια. Περνάμε λοιπόν στην ώρα της ψηφοφορίας. Και θα πρότεινα να αρχίσουμε αμέσως με την ψηφοφορία για τα σχέδια που μας παρουσίασε η κυρία Ματέρα. Το σημείο δηλαδή 19 και το σημείο 20. Έχει το κατάλογο στις ψηφοφορίες με δύο τροπολογίες. Για την πρώτη τροπολογία των κυρίων Αλβάρο και Άγγλοντ ο οποίος κ. το έφυγε, ούτε και ο Η συγκίτρια είναι υπέρ. συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, η συγκίτρια είναι υπέρ τη τροπολογίας υπέρ του είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Ποιο είναι κατά. Ε, ευχαριστώ. αποχέ. εγκρίνεται. Η ανθρωπολογία 2, η συγκίτρια είναι κατά όμω. Ποιο είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ, αποχές. Ωραία. Είναι κάπως απομονωμένος ο κύριος Άγγλοντ. Εγώ δεν συμμετείχα στην ψηφοφορία για να μην μείνει τελείως μόνος του. Λοιπόν. Θα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα στο σύνολο του κειμένου. Για το σύνολο του κειμένου. Δεν τα σημεία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία ψήφος κατά. Μία αποχή. Εγκρίνονται. Ευχαριστώ και με την εισηγητριά μας, κυρία Ματέρα. Ωραία. Τώρα, πάντα στην ώρα της ψηφοφορίας, ερχόμαστε στο διευθυντικό προπολογισμό υπαριθμών 9. που πρέπει να συζητηθεί μαζί με το σημείο 19. 17, συγγνώμη. 17. Που αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Λίγκης για δύο χώρες, την Πορτογαλία και τη Γαλλία. Ε, συγητής, κύριος Λάσος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Μπέγκιανα και να φύγει και μου επέτρεψε όμως να σας αναφέρω ότι υποστηρίζει την πρόταση και εγώ το ίδιο όσον αφορά τις δημιουργικές επιπτώσεις. Υπάρχουν βέβαια κάποια προβλήματα που πρέπει να σας αφαίρω. Πρέπει να υπερψηφίσουμε το θέμα από την άλλη μεριά θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε όσον αφορά τις πηγές των κονδυλίων αυτών που προτείνει η Κομισιόν. Θυμηθείτε πόσο δύσκολο ήταν το περασμένο έτος να έχουμε για το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης να βρούμε κάποια χρήματα. Και τα χρήματα αυτά είχαμε πει χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς στόχους και γι' αυτό δεν βρίσκαμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε. Καμιά φορά λοιπόν αυτές οι προτάσεις κομισιών να δημιουργηθούν νέα ταμεία, νέες δυνατότητες τέλο πάντων, δεν δικαιολογούνται απόλυτα αργότερα. Και γι' αυτό ε, εδώ τέλο πάντων μόνο το δεχθούμε γιατί είναι χαμηλό το ποσό. Λέγεται. Ε, δεν πρέπει όμως να αγνοούμε τις δυσκολίες ε, των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Λοιπόν, θα πρέπει ή να έχουμε καλύτερη δαπάνη ή καλύτερο προγραμματισμό στο μέλλον. Πάντως, σε γενικές γραμμές υποστηρίζω και τις δύο προτάσεις και ζητώ από την Επιτροπή μας να υπερψηφίσει. Πολύ ωραία, ευχαριστώ τον εισηγητή. Λοιπόν, εσείς αναφερθήκατε και στη χρηματοδοτική και στη νομική πτυχή που ήταν ο εισηγητής ο Μπέργκερ αλλά δεν θέλει κανένα το λόγο. Έχουν κάνει δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν είδα το Γενικό Διευθυντή του προπολισμού της Κομισιόν που ήρθε στην αίθουσα. Παρέσεις ήτανε. Ah Α, ξαναβγήκε. Α, ναι, ναι. C'est dommage, parce que il aurait pu voir... Κρίμα όμως. Γιατί θα μπορούσε να δει ότι η Επιτροπή Προπολογισμών συνεχίζει που και που να εγκρίνει προπολογισμού. Για να είμαστε σοβαροί όμως βλέπω ότι το Συμβούλιο που έχει πολλές ανα... αναζητήσεις νομικές, μεταφυσικές κλπ. Δεν έχει ακόμα επιλύσει οριστικά το θέμα που θα έπρεπε να έχει τεθεί της παρέμβασης των Εθνικών Κοινοβουλίων στις μουσουλμικές διαδικασίες βάσει του πρωτοκόλλου υπαριθμών 1 που έχει προστατευτεί στη συνθήκη της Σαββόνας όσον αφορά το έγκαιρο σύστημα προειδοποίησης, το Early Warning System. Και θέλει πάντα το θέμα κατά πόσον το Συμβούλιο θα χάσει άλλες 8 εβδομάδες για να ζητήσει την άποψη των 27 εθνικών κοινοβουλίων και των 40 νομοθετικών σωμάτων που υπάρχουν στα διάφορα κράτη για να δει κατά πόσο θα πρέπει να δοθεί μια κατυπήγουσα ενίσχυση στην Πορτογαλία. Ή στη Γαλλία και αύριο θα είναι κάποιες άλλε χώρε τέλος πάντων. Σούμα ιντζούρια λέμε. Δηλαδή, αν φτάσουμε στα άκρα της δικαιοσύνης φτάνουμε στα άκρα της αδικίας. La tue et l'esprit vivifie. Όπως λέει και η βίβλος, το γράμμα σκοτώνει, το πνεύμα αναζωγώνει. Βέβαια, έχουμε κάποιους μικρούς διαφορετικούς προπολισμούς. Εντάξει, αλλά θα πρέπει να δούμε το θέμα της έγκριση του προπολισμού 2001 το νέο σχέδιο προπολισμού δηλαδή που θα μας υποβάλει η ε, Επιτροπή. Μια που επέτυχε στην διαλλαγή. Θα πρέπει λοιπόν το Συμβούλιο να δει κατά πόσον θα θελήσει το Συμβούλιο να ακολουθήσει τη διαδικασία αυτή και να έχει μια συμπραγματική καθυστέρηση 8 εβδομάδων. Λοιπόν, εποφελούμενος από τις παρατηρήσεις αυτές, θα υποβάλω τώρα σε κοινή ψήφο τα σημεία 16 και 17. Ποιος είναι υπέρ. Χριστό κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Λοιπόν, τα δύο αυτά και κείμενα κινητοποίησης για δύο χώρες που βρίσκονται δυσκολίε έχουν εγκριθεί. Λοιπόν, κατόπιν Έχουμε το σημείο 19. 21, συγγνώμη. Που αφορά μεταφορές πιστώσεων. Ο εισηγητής. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από ό,τι μου λένε, αν είναι σωστές οι πληροφορίες, Υπάρχουν δύο προτάσεις που θα πρέπει να ψηφίσουμε και μπορούμε να ψηφίσουμε την υποστήριξή μου. Αν δεν κάνω λάθος, οι 37 και 38 αφορούν τη Σλοβενία και τη Γερμανία. Υπάρχουν άλλα που θα ψηφιστούν όμως στην επόμενη συνεδρίασή μας. Μία πρόταση πολύ επίμαχη, η οποία απαιτεί διευκρίνηση. Η 58. Παλιά ιστορία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω έχουν κάπου διαθέσει 4 εκατομμύρια ευρώ σε μια δράση για υποστήριξη τράπεζας που δεν είναι πολύ ξεκάθαρη. Κατέρευσε η τράπεζα και έχουμε απόφαση understand a lot of things for Έχουμε δικαστική απόφαση, αλλά δεν καταλαβαίνω με τι πραγματικές που διαθέτω ε, εδώ η διατύπωση τι σημαίνει. Προσπάθησα να μάθω και να καταλάβω, αλλά χρειάζομαι νομικές διευκρινήσεις για να μπορέσω να καταλάβω τι συνέβη και γιατί έπρεπε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μέσω μεταφοράς. Δεν είμαι έτοιμος να ψηφίσω λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Καλώς, ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Σαφές. Euh, ε, ψηφίζουμε λοιπόν μόνο για τις μεταφορές υπαριθμών 37 και 38 που αντιστοιχούν σε συμπλήρωση χρηματοδότηση στις δύο δράσεις που αναφέραμε προηγουμένως. Δηλαδή ομού θα ψηφιστούν έτσι. Ψήφι υπέρ παρακαλώ των μεταφορών αυτών πιστώσεων. Ευχαριστώ. Κατά. Δύο ψήφοι κατά. Δεν ξέρατε τι ήτανε, κύριε... Yes. If in doubt, vote no. <laughs> Αν ξέρατε, θα ψηφίζατε όχι. Ευχαριστώ. Αποχές εγκρίνονται λοιπόν. Τώρα, για τον προβληματισμό του κυρίου Σούριαν. Μήπως θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να απαντάει προφορικά σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω εδώ μαζί μου ένα συνάδελφο που είναι διευθυντής στο λογιστήριο ε, για αυτό το θέμα του προπολογισμού έχει παρακολουθήσει συγκεκριμένη υπόθεση που είναι και περίπλοκη και μπορεί να δώσει κάποια επισηματικά στοιχεία για να βοηθήσει ε, στην κατανόηση. Αν επιτρέπετε να του δώσετε το λόγο. Παρακαλώ κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε και αγαπητή δεν είχα την ευκαιρία ε, να εξηγήσω αυτά όπως τα εξήγησε ο ίδιος ο εισηγητής. Αυτή είναι μια υπόθεση που ξεκινάει από το 1998 για μια πληρωμή που είχε γίνει τότε σε μια μη κυβερνητική οργάνωση που εργοζόταν εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προ... Έγιναν οι πληρωμές κανονικά και μετά τρεις τελευταίες δεν έφτασαν στην τράπεζα του δικαιούχου. The amount, in fact, is a total και συνολικά είναι 3 εκατομμύρια ευρώ τα ποσά αυτά. Αμέσως, μόλις το μάθαμε, και το μάθαμε γρήγορα γιατί ο δικαιούχος δεν έλαβε τα κονδύλια αυτά, αυτό ε, ήδη από τότε έγινε μεγάλο πρόβλημα για τις υπηρεσίες. Η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, γνωμοδότησε μέσα σε 1,5 μήνα και ένα γραφείο δικηγορικό που ασχολείται με τέτοιες διεθνείς ε, τραπεζικές πληρωμές μας είπε ότι είχαμε πολύ καλή περίπτωση και πολύ καλά στοιχεία για ανάκτηση όλων αυτών των πιστώσεων και αμέσως δόθηκε αντίστοιχο ένταλμα. Ακολούθησε και δεύτερη πληρωμή. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι ε, ο δικαιούχος δεν είχε λάβει χρήματα. Έγινε μια δεύτερη ε, πληρωμή την οποία έλαβε ο, ο ενδιαφερόμενος. Ε, στη συνέχεια ακολούθησε και τρίτη εκτός προϋπολογισμού στον ισολογισμό. Το ε, επόμενο διάστημα συναντήθηκαν νομικές υπηρεσίες με την τράπεζα η οποία συμφώνησε να επιστρέψει τα χρήματα και αρχές του 1999 άλλαξε άποψη ριζικά η τράπεζα και επί σειρά ετών Είχαμε ανταλλαγή αλληλογραφίας ε, και ζητούσαμε ε, ανακαταβολή των χρημάτων. Πέρασαν πολλά χρόνια και τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσέφυγε σε δικαστήριο των Βρυξελών που ήταν αρμόδιο και δυστυχώς χάσαμε. Λόγω νομικού σφάλματος. Ακυρώθηκε η δεύτερη εντολή ε, ανάκτηση των τριών εκατομμυρίων, πράγμα που μας έκανε να καταβάλουμε τη δεύτερη δόση. Ε, το θέμα ήταν υποκαθάριση η τράπεζα και τα χρήματα έπεσαν σε μια μαύρη τρύπα. Και ε, τελικά έπρεπε όμως η τράπεζα να αποδείξει ότι είχαν ακολουθήσει τα χρήματα, το δρόμο τους μέχρι τον τελικό δικαιούχο. Δυστυχώς όμως το πρωτοδικείο των Βρυξελών είπε ότι τα τράπεζα τα έλαβε μία μεσάζουσα τράπεζα. Είναι γνωστή η υπόθεση, τα ξέρει ο εισηγητής, είναι δημόσια απόφαση του δικαστηριού, του πρωτοδικείου των Βρυξελών και επειδή συνέβησαν όλα αυτά, εμείς δεν μπορούσαμε να θεωρούμε ε, ε, υπεύθυνη ε, την Βελγική Τράπεζα ε, για την ανάκτηση των πόρων, γιατί είχαν ε, ε, εμβαστεί τα χρήματα σε άλλη ενδιάμεση τράπεζα και χάθηκαν. Στο μεταξύ είχαν φύγει από την Τράπεζα των Βρυξελών. Είναι λυπηρή, θλιβερή αυτή η περίπτωση. Εξαντλήσαμε τη διαδικασία. Τώρα προσπαθούμε να το βάλουμε στον προπολογισμό γιατί είναι στον ισολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλα αυτά τα χρόνια και μας ακολουθεί. Και τώρα θα πρέπει τα πληρώσουμε εμεί Τρία εκατομμύρια επιπλέον. Δηλαδή αυτό ήταν το λάθο στη δική μα κρίση. Εμεί θεωρήσαμε ότι είμαστε ε, σε καλό δρόμο, ότι θα παίρναμε όλα τα χρήματα πίσω, γι' αυτό προχωρήσαμε και στη δεύτερη δόση. Και αποφασίσαμε να μην κάνουμε και έφεση, γιατί είπαν οι εμπειρογνώμονε ότι θα χάσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα και προσπαθούσαμε να, χάσουμε, να κερδίσουμε μια υπόθεση που χάσαμε πρωτόδικα και που μάλλον δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πουθενά. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την ανάκτηση των πόρων για την αναμονή πόσο χρόνο περιμένουμε και τις εξωτερικές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και εν ώψη και της νέας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε τέτοιου είδους εκκρεμότητες από το παρελθόν. Ε, και θα δώσουμε συνέχεια μέχρι τέλους και ε, ε είχαμε και επιπτώσεις κάποιων ε, εργαζομένων που είχαν προκαταβάλει ε, κάποια ποσά για ταξίδια και τέτοια. Μπορώ να σας εξηγήσω διμερώς σε περισσότερες λεπτομέρειες και γιατί αν επιθυμείτε. Ευχαριστώ κύριε Διευθύντα για τις εξηγήσεις για τις δύο αυτές διαφορετικές μεταφορές. Το πρώτο είναι σαν αστυνομικό μυθιστόρημα, η πρώτη περίπτωση. Ο εισηγητής μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας, ούτως ώστε να δοθεί λογική συνέχεια στη δικαστική απόφαση και να γίνει η μεταφορά. Θα ψηφίσουμε αυτό το σημείο την επόμενη φορά και επί του άλλου σημείου θα ψηφίσουμε την επόμενη φορά. Αυτά για τι μεταφορέ που αφορούν τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τι άλλε κατηγορίε, άλλα θέματα, στρέφομαι προ τον Βλάδι Μάκα, τον άλλο εισηγητή, που έχει να παρουσιάσει τι μεταφορέ όσον αφορά το Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και το Ελεκτικό Συνέδριο. Ο κύριος Μάνκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τις μεταφορές αυτές, η πρώτη αφορά το ηλεκτρικό συνέδριο. Το ηλεκτρικό συνέδριο το 2004 είχε ζητήσει την εισαγωγή μέτρων όσον αφορά τις θέσεις Β και Α. Μια μεταφορά δηλαδή αυτών για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα. Ακριβώς αυτό τώρα πραγματοποιήθηκε και πριν οι νέες θέσεις α, β θα, θα μετατραπούν σε β, β. Αυτό δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση, γι' αυτό θα ήθελα να υπερψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όσον αφορά τη σε 11 τη μεταφορά. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ λοιπόν της πρώτης. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για την 47 ε, την τροπολογία. Εδώ το θέμα αφορά τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Δημιουργούνται ε, πρόκειται για τη μεταφορά προσωρινών θέσεων, δύο θέσεων άντε έξι προσωρινών σε δύο μόνιμες θέσεις άντε έξι Δεν αλλάζει τίποτα και θα ήθελα να υπερψηφίσουμε. Δεν υπάρχουν συνέπειες λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεν υπάρχουν άλλες μεταφορέ. Α, μία ακόμα. Κύριε Σιγητά. Ε, ναι, πρόκειται για μια, μεταφορά που αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ε, μεσοπρόθεσμη πολιτική ήταν, είχε ψηφιστεί να δημιουργηθούν κάποιες θέσει στο Στρασβούργο και στο Κοινοβούλιο για το διαδίκτυο. Η εισαγωγή του συστήματος αυτού θα κόστιζε 7,8 εκατομμύρια ευρώ. 3,8 στις ε, Βρυξέλλες και κάτι πάνω από 4 στο Στρασβούργο. Εδώ έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Βλέπετε, έχω εδώ τους υπολογιστές μου, δύο έχω και χωρίς ε, αυτούς δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Στο Στρασβούργο όμως είμαστε μόνο λίγες μέρες το χρόνο. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσο αυτά τα 4 εκατομμύρια ευρώ για το λειτουργικό κόστος 1-2 εκατομμύρια ευρώ και για τις δύο πόλεις είναι αποτελεσματική χρήση χρημάτων. Τα έγγραφα τα πήρα μόλις την Παρασκευή και απεδείχθηκε ότι δεν θα είναι πολύ απλά τα πράγματα. Συζήτησα και με τον κύριο Λαφορέ, τον Γενικό Διευθυντή Καινοτομίας και το ρώτησα το εξής αν θέλουμε αυτές τις συσκευέ να τις χρησιμοποιούμε και στο Στρασβούργο, θα πρέπει να έχουμε ε, κάποια εκτίμηση κόστους ωφελίας. Αυτό το έγγραφο δεν υπάρχει όμως μεταξύ εκείνων των εγγράφων που έλαβα. Ο κύριος Φαρέ τώρα μου τα έδωσε και αν είναι εδώ στην αίθουσα θα ήθελα να του δώσετε το λόγο πρόεδρο για να μας πει κάτι σχετικά με την αποτελεσματική χρήση αυτών των συσκευών. σε ευχαριστώ. Ο κύριος Γενικός Διευθυντής είναι εδώ. Α, συγγνώμη, δεν σας είχα Παρακαλώ, αυτό το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ε, υποστηρίζω πλήρως με τον εισηγητή. Στη συνέχεια όμως θα ήθελα να μου δώσετε το λόγο, σας παρακαλώ. Ή μήπως τώρα. Όχι. Τώρα θέλετε το λόγο ή μετά την απάντηση, μετά. Κύριε Γενική Διευθυντά. Αυτή, το αίτημα για τη μεταφορά πιστώσεων ε, έρχεται μετά από δύο αποφάσεις του Προεδρείου. Μια απόφαση που ζήτησε στη δική μας Γενική Διεύθυνση να κάνει πλήρη ε, μελέτη για την επέκταση του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη δεύτερη απόφαση ενέκρινε και, στο και στην Ολομέλη αυτό. Τα πλεονεκτήματα είναι και οικονομικά και η καλή χρήση των τεχνολογιών από πλευράς οικονομικής. Είναι προφανές ότι οι ε, κινητές τεχνολογίες έχουν ε, προχωρήσει με αλματώδη ταχύτητα και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα χρήσης ε, εντός του κτηρίου και γύρω από το κτίριο αυτή τη δυνατότητα. Τώρα, το roaming για ε, το mail σας ε, ή οτιδήποτε άλλο ε, είναι πάρα πολύ ψηλό. Γι' αυτό στην αρχή θεωρήθηκε ότι οι βουλευτές θα πρέπει να έχουν ασύρματο διαδίκτυο και στους διαδρόμους, δηλαδή να έχουν πρόσβαση από τα γραφεία τους. Επίσης, κάτι πολύ νέο, πίνακες τύπου iPad, μέχρι το επόμενο έτος θα έχουμε μία δεκαριά, αλλά δεν θα μπορούν να συνδέονται άμεσα. Ε, μάλλον θα συνδέονται άμεσα σε ένα δίκτυο και θα έχουν και ασύρματο διαδίκτυο. Και μια άλλη σκέψη που είναι και στόχος του Κοινοβουλίου είναι ε, για την περιβαλλοντική διαχείριση έμας για λιγότερο χαρτί στο Κοινοβούλιο. Και αυτό δεν αφορά μόνο ε, την περίπτωση αυτή υπάρχει ένα πρόγραμμα έτσι ώστε όλα τα έγγραφα των κοινοβουλευτικών επιτροπών να είναι προσβάσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. Στο device, στα αγγλικά το λένε αυτό, ε, σε ό,τι μηχάνημα θέλετε, Λάπτοπ, εφίες τηλέφωνο, smartphone ή ε, υπολογιστή. Αρχές του επομένου έτους θα γίνουν όλα αυτά. Αλλά για να γίνουν, ε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάλυψη ασύρματη παντού. Αυτό ισχύει και για το Στρασβούργο. Έχουμε όλες τις συνεδριάσεις των ομάδων, την Ολομέλεια στο Στρασβούργο, μία συνεδρίαση ομάδα την ημέρα. Αυτό το ασύρματο δίκτυο λοιπόν θα βοηθάει και θα είναι στην υπηρεσία όχι μόνο των βουλευτών των μεμονωμένων αλλά και ε, ε, των πολιτικών ομάδων αλλά και των πολιτών που είναι όλο και περισσότεροι στο κοινοβούλιο μας. Από πλευράς κόστους γνωρίζετε το σύστημα Elvis στις δύο ολομέλειες. Ε, ξέρετε τις οθόνε που δίνουν ε, σχετικά σύντομες ε, πληροφορίες για τη ροή της ολομέλειας. Ομιλητές και εισηγητές και ψηφοφορίες. Εάν θέλουμε αυτό το σύστημα να το επεκτείνουμε σε όλες τις συνεδριάσεις, αυτό θα σήμαινε από πλευρά υποδομής ότι όλες οι αίθουσες συνεδριάσεων θα πρέπει να έχουν οθόνες και οθόνες αφής. Πράγμα που σημαίνει ε, πολύ μεγαλύτερη ενέργεια σε κάθε έδρανο μπροστά. Ένα λαν σε κάθε έδρανο. Συν... Chaleur ε, και επίση, ξέρετε, ε, ότι ε, εκπέμπουν και θερμότητα ε, αυτές οι μηχανές, αυτά τα μηχανήματα και χρειάζεται και ψήξη σε ορισμένες αίθουσες, δηλαδή κλιματισμός. Και είναι το κόστος απαγορευτικό σύμφωνα με τις υπηρεσίες μας. Υπολογίσαμε ότι σε μία και μόνο αίθουσα μια τέτοια οθόνη θα σήμαινε το εξή, γιατί και τα DexMem χρειάζονται ειδικό configuration. 4.000 ευρώ ανά οθόνη παρακαλώ. Άρα για 30 αίθουσε εκτό από το ημικύκλιο έχουμε 41 εκατομμύρια ευρώ. Je considère que ce choix Βρυξέλλες και Στρασβούργο εννοείται. Ε, είναι το κόστος αυτό, ένα κόστος ε, σκόπιμο για το Κοινοβούλιο, ακροπρόθεσμη ε, επένδυση, ε, απαντά στην ευελιξία των βουλευτών που το επιθυμούν και είναι ένα επιχείρημα και τεχνικό και πολιτικό. Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθύντα. Ο Λάσλο Σούριαν. Thank this... Ευχαριστώ. Μετά τις εξηγήσεις αυτές Είμαι πρόθυμος να υποστηρίξω την αρχική πρόταση, ιδιαίτερα τώρα που έμαθα ότι θα έχουμε κάποιες δυσκολίες για το προπολογισμό του 2011. Αν αναβάλουμε ε, την απόφαση αυτή, ένας Θεός ξέρει πότε θα μπορέσουμε να την λάβουμε, αν την αναβάλουμε τώρα. Παρακαλώ τους συνεισηγητές να δείξουν κάποια ευελιξία. Εγώ Έχω πολλές δυσκολίες στο Στρασβούργο, ιδιαίτερα όταν έχω ασκούμενους μαζί μου, οι οποίοι έχουν τους υπολογιστές, ε, το, τους ασύρματους και ένα καλώδιο μόνο. Και ένα τόσο μικρό γραφείο, τουλάχιστον να μια καρέκλα και ο καθένα στα γόνατά του να έχει το λάπτοπ και να μπορεί να δουλεύει, έστω και χωρί καλώδια. Είναι πολύ λογικά αυτά που ακούμε. Euh, Σας ευχαριστώ. Ο Χάρτον έχει το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρα από το γεγονός ότι θα γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έχει ο κάθε βουλευτής το λάπτοπ του και θα συνεχίζει η συνεδρίαση. Γιατί λέμε να νοικιάσουμε εξωτερικούς βοηθούς outside assistance, δεν έχουμε ε, εμπειρογνωμοσύνη εμείς στο Κοινοβούλιο, στη δική μας υπηρεσία τεχνολογιών και τι θα γίνει με την ανάθεση και με τους ε, διαγωνισμούς σε περίπτωση που προχωρήσει βέβαια αυτό το έργο. Πώς θα πάει η διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα απαντήσει ο Γενικός Διευθυντής. Ο κύριος Φερνάνδος έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι πάντα είμαστε υπέρ της ε, ε, νομοθεσίας υψής του επίπεδου και της παραγωγικότητας και θα πρέπει να έχουν ε, οι βουλευτές τα αναγκαία μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μετά την εξαντλητική απάντηση που δόθηκε από τον κύριο Γενικό Διευθυντή δεν έχω ούτε μία αμφιβολία ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία η οποία πάνω απ' όλα υποστηρίζει την παραγωγικότητα Και η παραγωγικότητα αυτή μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους 20-20-20 της Ευρώπης όσον αφορά τις εξοικονομήσεις ενέργειας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, θέλετε να απαντήσετε στο δεύτερο ερώτημα του κύριου Χάρτουγκ. Η πρώτη αφορούσε, νομίζω, το κόστος του project management. Είναι ένα θέμα τεράστιο, τεράστιο εγχείρημα που υποχρεώνει την εταιρεία ε, να εργάζεται εκεί, τις νύχτες, τους διαδρόμους, ή συνεδριάσει των επιτροπών όταν δεν υπάρχει συνεδρίαση. Για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, που σημαίνει ότι πρέπει να φυγούν οι οροφές από τους διαδρόμους, ε, δεν μπορώ να βασιστώ μόνο στους υπαλλήλου. Θα είναι υπό τον έλεγχο των υπαλλήλων, αλλά χρειάστηκε βοήθεια όσον αφορά την παρακολούθηση του έργου για τόσο σημαντικό εγχείρημα. Όσον αφορά τις τιμές, είναι αποτελέσματα πρόσκληση υποβολής προσφορών και υπάρχουν, έχουν γίνει προσφορές, δημόσιος διαγωνισμός. Και κρατήσατε, ας πούμε, τα χαμηλότερες τιμές, τις καλύτερες προσφορές, απάντηση. Έγινε πρόσκληση υποβολής προσφορών, αυτό μας επέτρεψε ο διαγωνισμός να αγοράσουμε, μας επιτρέπει να αγοράσουμε υλικό υλικό που κατασκευάστηκε το 2005 και είναι μια σύμβαση πλαίσιο αυτή που επιτρέπει ευελιξία για να αγοράσουμε υλικό που θέλουμε να αποκτήσουμε. Ήταν δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός. Και υπάρχει, έγινε αυτό, αλλιώς δεν θα κάναμε την πρόταση. Καλώς, σας ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά, ποια είναι η άποψή σας να εγκρίνουμε αυτή την πρόταση μεταφοράς. Ναι. Ευχαριστώ για τις εξηγήσει. Θα ήθελα να πω στον κύριο Σούριαν ότι είναι δεδομένη η δική μου ευελιξία. Είμαι αρκετά ευέλικτο. Υπήρχαν ορισμένα ερωτηματικά και ανοιχτά ζητήματα θα πρέπει να δούμε και την αποτελεσματικότητα, ε, τη σκοπιμότητα ε, του σχεδίου μας απάντησε ο Γενικός Διευθυντής και μπορούμε να τα έχουμε ως επιχειρήματα αυτά για να απαντούμε σε κάθε ερώτημα και σε κάθε πρόβλημα για να μπορούν οι βουλευτές να εργάζονται σωστά και να αποφασίσουν μετά λόγου γνώσεως και τα καλώδια που θα τοποθετηθούν είναι μέτρα, χιλιόμετρα ολόκληρα. Εγώ δεν αμφισβητώ καθόλου ούτε έχω τέτοια πρόθεση το ποσό. Αλλά ο χρόνος που δαπανούμε στο Στρασβούργο είναι πολύ περιορισμένος. Γι' αυτό με προβληματίζει αν είναι σκόπιμο στο Στρασβούργο να ε, στήσουμε ολόκληρο τέτοιο σύστημα. Ε, θα είχαμε και μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων αν μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε το ασύρματο ε, διαδίκτυο και για τηλεφωνήματα, για παράδειγμα. Παρακαλώ λοιπόν να υπερψηφίσουμε ε, την πρόταση. Σας ευχαριστώ. Εξορισμού μία φορά, μία εβδομάδα το μήνα είμαστε στο Στρασβούργο. Άρα θέλουμε να δούμε αν θα έχουμε τα μέσα να δουλέψουμε αυτή τη βδομάδα ή όχι. Νομίζω ότι είμαστε πλήρως ενήμεροι και ψηφίζουμε. Ο εισηγητής σας, μέσω των παρατηρήσεων που έκανε, είναι υπέρ αυτού. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς. Κατά. Δύο αποχές. Η μεταφορά αυτή εγκρίνεται λοιπόν. Κύριε εισηγητά, κύριε Μάκα, δεν υπάρχει άλλη μεταφορά. Ωραία, πολύ καλά. Σας ευχαριστώ. Μας απομένει το τελευταίο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης. Α, όχι, συγγνώμη. Κύριε Σούριαν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ζήτησε να έρθω σε επαφή μαζί της και θέλω να σας ενημερώσω. Είναι μακρύς ο κατάλογος των μεταφορών πιστώσεων που αναβάλουμε κυρίως ό,τι αφορά το Ταμείο Καταπολέμησης Παγκοσμιοποίησης και χωρίς την κυρία Ματέρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και δεν θα αναφερθώ σε αυτό, αλλά το αίτημα είναι το εξή. τεσσερις Τέσσερις-πέντε άλλες μεταφορές πιστώσεων που συζητήσαμε αυτό το θέμα της τράπεζας προηγουμένως, έτσι κι αλλιώς ε, θα πρέπει να το λύσουμε, αλλά και κάτι άλλο. Η γραμματεία Δεν είναι έτοιμοι να ψηφίσουμε τα υπόλοιπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα αίτημα λοιπόν προς ένα ερώτημα. Αν μπορούμε να ψηφίσουμε την άλλη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Δεν βλέπω να έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών στο Στρασβούργο. Και θα ήταν πολύ περίεργο και η προγραμματισμένη μας ε, συνεδρίαση είναι την 1η Δεκεμβρίου. Αν βιάζονται τόσο πολύ, γιατί το βάλαν στις 5 Νοεμβρίου και το ζητούν τώρα να συζητηθεί και να ψηφιστεί. Αυτή την ε, αίτηση, αυτό το αίτημα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί έχουμε κάθε πρόθεση να του ικανοποιήσουμε, είναι και εγκρέσλη αυτού. Υποθέτω ότι το δέκ 61 ε, εμπίπτει στις ίδιες πιστώσεις που ήθελε ο Λάσλο να αναβληθούν. Γιατί θέλω να πω για τον 1061 αυτό το αίτημα δεν είναι απλώς μια μικρή μεταφορά, αλλά είναι ε, αναδιάρθρωση ολόκληρη της γραμμής αυτής του προπολογισμού, της πίστοσης. Ότι οι χώρες ε, υποψήφιες προενταξιακές δηλαδή θεωρούνται κράτη-μέλη ούτε λίγο ούτε πολύ και χρηματοδοτούνται. Και αυτό ε, είναι κάτι το οποίο κάνει το προπολογισμό μας ακόμα λιγότερο διαφανή και ορατό. Πώς το φαντάζεται αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην απαλλαγή τι θα κάνουμε, θα μας δώσουν τα ποσά, τα αθροίσματα, το σύνολο και δεν θα ε, ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν θα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Θα πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζεται ο προπολογισμό και ε, να ζητήσουμε τι μεταφορέ πιστώσεων. Θέλουμε προπολογισμό που να μην ξέρουμε καθόλου που πηγαίνουν τα χρήματα. Να έχουμε ένα μεγάλο κορβανά και ο καθένα να μπορεί να παίρνει τα χρήματα και να τα μεταφέρει προ την κατεύθυνση που χρειάζεται ακριβώ εκείνη τη στιγμή. Ε, δεν ξέρω, με προβληματίζει πάρα πολύ αυτή η υπόθεση και δεν μου αρέσει καθόλου. Ωραία. Η κυρία Γκρέσλα απάντησε στο ερώτημα του κυρίου Σούριαν. Δεν είμαστε σε θέση να προβούμε σε αυτή τη μεταφορά. Μου λέγουν ότι νομικός πρέπει να περιμένουμε το μήνα Δεκέμβριο. Στην επόμενη συνεδρίασή μας θα είμαστε εδώ μία και δύο Δεκεμβρίου. Ίσως έχουμε έκτακτη συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα. Θα μιλούσα σε λίγο γι' αυτό. Αλλά όχι να την αφιερώσουμε όσο και σημαντική είναι η μεταφορά σε μια μεταφορά. Τέλο των ψηφοφοριών όσον αφορά τι μεταφορέ. Μπορούμε να, έχουμε τη Μόνικα ε, Χολμάιερ που θα μιλήσει για τον Νίγηρα. Να ξεκινήσουμε αυτό το θέμα. Η κυρία Χολμάιερ έχει το λόγο για να μα πάει στον Νίγηρα. Ναι. Ε, εύκολο θέμα ο Νίγηρας. Το, τα... ταξίδι είναι εύκολο, η χώρα δεν είναι. Πρόκειται αγαπητοί συναδελφοί για ένα οικόποδο που προβλέπεται για την ε, οικοδόμηση του νέου κτηρίου της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ήγερα. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι μέχρι στιγμή είχαμε κάποια γραφεία στο δεύτερο και τρίτο ε, όροφο μιας ε, τράπεζας. Τράπεζα Πολαφρίκ στον Ήγηρα. Έχουμε προβλήματα με την επιφάνεια, 48 εργάτες. αλλά υπάρχουν θέματα ασφαλείας, γιατί η τράπεζα αυτά, αυτή είναι ανοιχτή στο δημόσιο και βέβαια όσον αφορά την τρομοκρατία είναι κάπως επικίνδυνα τα πράγματα και αυτό η Κομισιόν προσπάθησε να βρει άλλες δυνατότητες. Έχω κάποια κάθε κατανόηση γιατί ξέρουμε ότι οι συνεργάτες μας σε ορισμένα μέρη του κόσμου ε, ζουν επικίνδυνα. Γι' αυτό προβλέπετε να αγοραστεί ένα οικόπεδο που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κτίρια πρεσβειών πολύ καλά ασφαλισμένη δηλαδή η περιοχή που δεν είναι δημόσια η πρόσβαση και οπωσδήποτε οι συνεργάτε μας θα είναι εκεί πέρα πολύ πιο ασφαλείς από ότι στο κτίριο αυτό που είναι ανοιχτό για το κοινό όπως σας είπα και που δεν είναι δυνατόν να οριοθετηθεί και που δεν υπάρχουν και ειδικά μέτρα ασφαλείας γύρω από το κτίριο. Τώρα, έχουμε 1.017.000 ε, η τιμή του οικοπαίδου θα πληρωθεί ε, σε δύο δόσεις το 2010 και το 2011. Ε, το κτίριο αυτό α, ανήκει στην Γαλλία από ό,τι ξέρω που θα μας το δώσει σε μια καλή τιμή και ένα πολύ καλό οικόπεδο και ελπίζω να δώσουμε την άδειά μας να μπορέσει η Κομισιόν να αγοράσει αυτό το, το οικόπεδο. Ευχαριστώ. Αυτό τι σημαίνει κυρία Συγγετρία. Βρισκόμαστε στις διαβουλεύσεις του άρθρου 179. Η σύστασή σας είναι λοιπόν να μην γνωμοδοτήσουμε. Μάλιστα λέει η Συγγετρία. Ωραία. Ο κ. Σάτουμ τι το λόγο. Πρόεδρε, θα παρακαλούσα εξ ονόμα της Επιτροπής μας να ζητήσουμε μια επίσημη γνώμη. Το σημειώνω. Λοιπόν, να ψηφίσουμε. Η ε, κυρία Μία ερώτηση, πρόεδρε. Ακούγοντα αυτά που είπε, γιατί θέλουμε να φύγουμε από το κτίριο τη τράπεζα, γιατί δεν είναι αρκετά ασφαλέ. Και τώρα θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα φρούριο, αν μπορώ να το πω έτσι, στον Ήγερα. Το θέμα όμως αυτό που φαναζόμαστε εμείς, ότι οι αντιπροσωπείες θα πρέπει να είναι και εκείνες που παρουσιάζουν την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα πρόσβασης του κοινού. Δεν επιθυμούμε κάτι τέτοιο. Α, εντάξει. Γιατί είχατε εντύπωση πραγματικά... Όχι, όχι. Δεν είναι όπως η Σόφια βέβαια, όπου είμαστε μέσα στην ε, Βρετανική Υπηρεσβεία και όποιος θέλει να πάρει και ένα φυλάδιο περνάει από σωματικό έλεγχο. Όχι, το κτίριο θα είναι προσβατό, αλλά δεν θα είναι έτσι μέσα στη μέση της πόλης ανεξέλεκτο και θα πρέπει επίσης όπως και σε άλλα κτίρια να εξτάσουμε το θέμα κλιματισμού. Εκεί έχουμε παραδείγματο χάρη πάρα πολύ θόρυβο από το έξω. Έχουμε ορισμένου που εργάζονται σε χώρους που δεν έχουν φω ημέρα. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε για τι συνεργάσει μα. Όχι φρούριο πάντω. Αλλά μια που υπάρχουν και πρεσβείες δεξιά και αριστερά, υπάρχει περισσότερη αστυνομία αστυνομία, περισσότερη ασφάλεια. Φυσικά είναι καλό το από το κοινό, αλλά σε πιο ασφαλές περιβάλλον. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Είναι. Και θέλω να παρατηρούμε τη συζήτηση, αλλά η ερώτηση της Γιούτα καλή ήταν. Γιατί τώρα έχουμε μία σειρά αγορών στον τομέα εξωτερικών σχέσεων και θα ήταν καλό εάν η νέα υπηρεσία εξωτερικών δράσεων μπορέσει να μας δώσει μια εικόνα το ποια συνειδητότητες που υπάρχουν, ποια τακτήρια που υπάρχουν, τι μέτρα ασφαλείας υπάρχουν. Η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήταν λοιπόν καλό να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσουν αυτές οι 140 ε, εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο. Ωραία, Λέα ο σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ζητήσουμε το Μισό να μας απαντήσει για το γενικό αυτό πρόβλημα την επόμενη εβδομάδα. Δα και βέβαια δεν έχουμε και δεν είναι πολύ επίγον γιατί καθυστερούμε έτσι και αλλιώς την υιοθέτηση του προπολογισμού και έτσι οι περισσότερες εξωτερικέ δράσει δεν θα τεθούν σε ισχύ παρά μετά από πολλές εβδομάδε. Τώρα, για τον Ήγρα εγώ θα σα έλεγα αν η Γαλλία σα δίνει ένα οικόπεδο πρέπει να το αρπάξετε. Γιατί, ξέρεις, ο Νίγερα μπορεί να έχει ουράνιο στο υπέδαφος. <laughs> Ευκαιρία είναι, να στο αγοράσουμε γλίγορα. Πρόεδρε, αν βρούμε ουράνιο ή οτιδήποτε πετρέλαιο ή θα το βρούμε και κάτω από τη γαλλική πρεσβεία που είναι δίπλα ακριβώς. Θαυμάσια. Λοιπόν, πολύ σημαντική παρατήρηση βέβαια. Η συγχύτρια προτείνει να μην γνωμοδοτήσουμε. Ο κύριο Χάρντον θέλει όμω να γνωμοδοτήσουμε. Ποιο ακολουθεί την πρόταση τη συγχύτρια, παρακαλώ, να μην γνωμοδοτήσουμε. Ευχαριστώ. Ποιο είναι κατά. Δύο. Αποχές. Ωραία. Λοιπόν, θα αφήσουμε το τρένο να περάσει μπροστά μας ανενόχλητο. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο θέμα, όσον αφορά την δημοσιονομική συζήτηση, σας ανακοινώνω ότι ζήτησα από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να μας Ah pardon, ben alors je vous en prie, je Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Με συγχωρείτε πως σας διακόπτω, αλλά προχωρήστε πολύ γρήγορα. Υπάρχει ο λόγος γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Γιατί για το κτίριο υπάρχουν διάφορα προβλήματα συγκεκριμένα. Το ένα αφορά την ουδετερότητα επιφάνειας. Δηλαδή εγκαταλείπουν 38.000 τετραγωνικά και θα πρόκειται να χρησιμοποιήσουν 46.000. Από τις 18.000, 18.000 περίπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για τις άλλες 20.000 από ό,τι ακούσαμε, η Κομισιόν έχει ένα πρόβλημα στενότητας χώρου και εγώ λέω ότι βέβαια οι βουλευτέ έχουν μεγαλύτερη στενότητα χώρο από ό,τι είχε ποτέ η Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι ο προπολογισμό δεν είναι και τόσο ανοιχτό που να μπορούμε να έχουμε γενοδορία Και είχαμε πει πάντα ότι θα πρέπει να έχουμε μια ουδετερότητα τη κάλυψη και γι' αυτό εδώ έχω κάποια ερωτηματικά. Το δεύτερο είναι το θέμα τη ουδετερότητα όχι τη επιφάνεια πια, αλλά τη δημοσιονομική. ιδίως για τα αριθμητικά στοιχεία, έχουμε κάποιες επερωτήσεις, μια που ορισμένα αριθμητικά στοιχεία δεν τα έχουμε ακόμα στα χέρια μας και η οργάνωση του κτηρίου δεν υπάρχει ακόμα. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει το κτίριο. Και θα ξέρουμε ποιο θα είναι το κόστος εκμύθιστοσης. Ε, και ποια θα είναι η τιμή αν αλλά το σύνολο του κόστους δεν είναι ακόμα γνωστό. Εκεί έχουμε μια επιρροσή. Τρίτον, το θέμα της ασφάλειας. Μπορεί να επιληθεί γιατί σε ορισμένα αυτά τα κτίρια ε, ε, υπάρχουν, ε, σούπερ μάρκετ στο κάτω μέρος και βέβαια όταν υπάρχει ε, σούπερ μάρκετ ε, δεν μπορεί κανένας να κάνει κανένα έλεγχο αλλά το κόστος αναφέρεται 3,3 εκατομμύρια. Εμένα μου είπανε μάλιστα ότι θα είναι πιο υψηλό. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρουμε τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία. Γιατί είναι καλό να ξέρουμε τι θα κοστίσει τελικά. Και το τρίτο θέμα είναι η νομική κατάσταση και έχουμε αποτυχία των δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων το 2011. Και άρα δεν έχει ακόμα ε, επιληθεί το ποια μορφή θα έχει η χρηματοδότηση γιατί υπάρχει η νομική βάση αλλά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής η δημοσιονομική βάση γιατί εδώ με τον προπολισμό είμαστε στα κατημόρια. Έκαναμε πρώτη συζήτηση ε, θα γίνουν και άλλες συζητήσεις δεν είμαι εξ αρχής αντίθετη αλλά υπάρχουν διάφορες επιρροτήσεις και η μια με ενόχλησε, δηλαδή υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένω το κτίριο Λέξε θα ήταν το πιο κατάλληλο το οποίο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί το Συμβούλιο. Γιατί εάν πρόκειται να χρησιμοποιεί για την υπηρεσία εξωτερική θα πρέπει να φύγουν όλοι οι μεταφραστές από εκεί και θα πρέπει να μεταποιηθεί το κτίριο κλπ. Και μου είπαν ότι θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει. Το Συμβούλιο όμω που μας είπε στι δημοσιονομικές διαπραγματεύσει ότι όλοι πρέπει να κάνουμε εξοικονομήσει, δεν θέλει να βάλει τους μεταφραστές του πουθενά αλλού. Λοιπόν, όταν εμάς μας καλούν να κάνουμε εξοικονομήσεις είναι πολύ δύσκολο να γίνουν οι συζητήσεις για συμπληρωματικό ο κόστος ε, στα πλαίσια του προπολογισμού από αγγλικής πλευράς. Εγώ ήθελα πρώτα να το αναφέρω γιατί μου το ανέφερα και εμένα δεν θέλω να το αποκρύψω ότι μου το είπαν αυτό. Και θα ήθελα και με τον Γενικό Διευθυντή και με τους συνεργάτες να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Να αναβάλουμε λοιπόν. Bien. Donc... Πολύ καλά. Θέλω να καταλάβω, δηλαδή από ό,τι είπατε, από την ανάλυση σας εδώ, αντίθετα από ό,τι έγινε με τον Ήγηρα, θέλετε να τοποθετηθούμε. Ναι, λέει η συγγήτρια και θέλω να αναβληθεί. Οπότε συμφωνούν όλοι. Ο κ. Χάρτουγκ δεν έχει αντίρρηση. Πω πω αξιοσημείωτο λέει η συγγήτρια. Θέλα, δεν ξέρω αν έχει πρόταση. Λοιπόν, ας με επιτρέψετε να προτείνω στην εισηγήτρια κάτι. Να έρθετε σε επαφή σύντομα με τους ε, αρμοδίους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε αυτό το θέμα να είναι όριμο για να τοποθετηθούμε εμείς σύμφωνα με το άρθρο 79 εντός των προθεσμίων προβλέπονται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Το συζητήσαμε, συζητήσαμε διάφορες πτυχές στα πλαίσια της δημιουργίας της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, τα συζητήσαμε αυτά τα σημεία. Χρειάζεται ένα κτίριο, χρειάζεται να το στεγάσουμε θα πρέπει να κοστίσει ένα λογικό ποσό, να μην υπάρχει ένα ασυνήθιστο ποσό που θα απαιτηθεί. Κυρία Άστον, εδώ και ένα ε, ε, χρόνο περνά γολγοθά. Πάντα αναφέρομαι στη βίβλο, είμαι χριστιανοδημοκράτης, βλέπετε. Αλλά δεν πρέπει να έχει πάνω από 12 σταθμούς ο Γολγοθάστης. Είναι στο 14ο, 14η στάση. Μια μικρή παράκληση μόνο. δεν ήταν βέβαιος ότι θα μπορούσε να τηρηθεί η προθεσμία για την απάντηση. Ε, εγώ δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα γίνει μέσα στο 15 μέρο. Χρειάζομαι κάποιες απαντήσεις, αλλιώς μπορεί η γνωμοδότηση να βγει αρνητική, γιατί δεν υπάρχουν αρκετές απαντήσεις. Δεν επιθυμώ κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως να χρειαστεί να το συζητήσουμε μήπως μπορεί να γίνει το Δεκέμβριο εγώ δεν είμαι αρνητικά διακείμενη ε, ε, καταρχήν, αλλά θέλω να δω μερικές διευκρινήσεις και να λυθούν ορισμένα πράγματα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ακούστηκε το μήνυμά σα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ για τη στάση σας που είναι και ανοιχτή και αυστηρή. Τελευταίο σημείο. Είμαι σε θέση να σας πω λοιπόν ότι η επόμενη συνεδρίαση τακτική 1η Δεκεμβρίου από 3 μέχρι 6.30 2 Δεκεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 επιφυλασσόμεθα της δυνατότητας διεξαγωγής εκτάκτου συνεδριάσεως εις Στρασβούργων που θα αφορά αποκλειστικά τις διαπραγματεύσεις του προπολογισμού την 3η 23 του μηνός μου λένε ότι τώρα έχουμε μια διευκρίνηση από τις 10 μέχρι τις 11.30 στην αίθουσα WIC 200. 216 θέσεις έχουμε εκεί και έχουμε δικαίωμα 18 γλωσσών, διερμηνίας σε 18 γλώσσες. Θα το επιβεβαιώσουμε μέσω email αυτό. Λοιπόν, διακόπτω τις εργασίες Καλό βράδυ. Γεια σας.